Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουμτσάκο και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Συνεχίζουμε και περνάμε σε άλλη γραπτή δήλωση 21 του 2011 των Γιέκο Κάτσιν, Έντβαρτ Μακμίλαν Σκότ, Αννα Ρόσβαχ, Γιώργη Σέπλιν και Γιούτα Στάινρουκ όσον αφορά τους άμαχους αναπήρους πολέμου και έχω υπογραφεί από τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάλι σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα στελεί στους ε, αποδέκτες και θα δημοσιευθεί επίσης τα πρακτικά. Τα ονόματα των υπογραφώντων την ε, δήλωση αυτή θα επισυνάπτονται επίσης στα πρακτικά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Vice President. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι εκ μέρου όλων εκείνων που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία. Σε ευχαριστώ ειλικρινά για την υποστήριξή σας. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που περνά μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ε, λόγω των πολέμων σημαδεύτηκαν από τον πόλεμο και από διάφορες βίες πράξεις και έχουν σημαδευτεί για όλη τη ζωή. Αυτή η δήλωση ετοιμάστηκε σε συνεργασία με διάφορες οργανώσεις από όλη την Ευρώπη αναπήρων πολέμου. 388 υπογραφές έχουμε μαζέψει και χαιρόμαστε που έχουμε ανάμεσά μας τους επικεφαλείς των τριών μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων. Δεν θέλω να πω ότι μετά από 7 χρόνια δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν η πρώτη φορά αυτή που παρατήρησα ότι όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες ή κάποια μέλη αυτού του Κοινοβουλίου για δικούς τους βασικούς λόγους δεν υπογράφουν γραπτές δηλώσεις, οποιαδήποτε γραπτή δήλωση. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ παράξενο, διότι οι γραπτές δηλώσεις είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε. Πρόεδρος, πάμε τώρα στη ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την έκθεση Μπερές, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, της κυρίας Μπερές, για την τροποποίηση του κανονισμού 1927 που δημιουργεί